Darf Παρακαλώ καθίστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζουμε με την ε, σύνοδο η οποία διακόπησε στις 4 Ιουλίου του 2013. Κυρίσω την έναρξη της συνεδρίασης. και θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην πρώτη μας σύνοδο της Ολομέλειας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Θα ξεκινήσω δυστυχώς με μια δυσάρεστη ε, είδηση. Ο συνάδελφος Λόταρ Βίτσκι ε, πέθανε απρόσμενα στις 13 Αυγούστου. Ο ξαφνικός του θάνατος ε,